Dear colleagues, good afternoon. May we start. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Θα ξεκινήσουμε ως ήθιστε με την έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Το σημείο 7 προτείνω να εξεταστεί μετά από το 10. Το 8 αναβάλλεται. Το 23 επίσης. Και το 27 θα το εξετάσουμε μετά το 13. Αντιρρήσεις δεν βλέπω. Για το σημείο 2, προ... ανακοινώσει του Προέδρου, δεν έχω να κάνω καμία ανακοίνωση σε αυτή τη φάση, οπότε προχωράμε κατευθείαν στο σημείο 3 για την ακρόαση για τη συνθήκη του Μαρακές. Επιτρέψατε μου να καλωσορίσω θερμά ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους προσκεκλημένους μας που δέχτηκαν την ε, πρόσκλησή μας να έρθουν και να μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία τους. Θα θέλαμε να σας ακούσουμε σχετικά με την προέλευση αυτής της συνθήκης του Μαρακές που θα διευκολύνει την πρόσβαση σε δημοσιευμένα έργα για τους τυφλούς και τους ανθρώπους με δυσκολίες στον έντυπο, στο έντυπο υλικό και θα μας εξηγήσετε γιατί είναι τόσο σημαντικό να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή εκτιμά τι δύο νομοθετικέ προτάσει που θα εντάξουν τη συνθήκη αυτή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και γι' αυτό θα θέλαμε να μα εξηγήσετε πώ μπορούν να ξεπεραστούν οι σχετικέ προκλήσει. και κυρίως στην φάση της εφαρμογής. Έχουμε περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας ζητήσω να μιλήσετε για 8 λεπτά ε, ο καθένας από εσάς. Επίση, θα ήθελα να καλωσορίσω τα μέλη των ε, Επιτροπών που για γνωμοδοτήσεις ε, και να σας καλέσω να συμμετέχετε στη συζήτηση. Θα ξεκινήσω λοιπόν αμέσως δίνοντας το λόγο στην κυρία Μαρία Μαρτίν Πράτ από την DG Connect για το πρώτο τμήμα της ε, δημόσιας ακρόσης που αφορά την προέλευση και τις διαπραγματεύσεις περί της συνθήκης για να μας εξηγήσει γιατί είναι σημαντική η συνθήκη του Μαρακές. eight minutes, please. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία στην Επιτροπή να συμμετέχουμε σε αυτήν την ακρόαση. Θέλατε Επιτροπή να αναφερθεί στην ε, προέλευση, στο ιστορικό και της ε, συνθήκης του Μαρακές. Θα ήθελα να συνοψίσω με το να πω ότι ήταν μακρές οι διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Ξέρετε ότι οι πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες για οποιοδήποτε ζήτημα συμπεριλαμβανομένων των, ε, πνευματικών δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο είναι συνήθως χρονοδόρο. Οι συζήτηση για την συνθήκη του Μαρακές ξεκίνησαν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Πνευματική Διοκτησία και ξεκίνησαν από το 2008-2009. Το 2009 ξεκίνησαν ουσιαστικά οι ε, διαπραγματεύσεις σοβαρά στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής ε, για τα πνευματικά δικαιώματα ε, για άτομα με αναπηρία και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μεγάλη προσπάθεια η οποία στην ουσία προωθήθηκε από τους ε, ε, δυνητικά εποφελούμενος από μια τέτοια συνθήκη. Ε, όπως είπαμε πήρε πολύ χρόνο και τελικά ψηφίστηκε αυτή η συνθήκη από οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τους τυφλούς σε διάφορες χώρες της Ευρώπης αλλά και εκτός Ευρώπης έγινε πραγματική συζήτηση όσον αφορά τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων και τις ε, καταστάσεις ε, που δικαιολογούσαν μια εξαίρεση σε, αυτή την, σε αυτόν τομέα. Χώρες όπως η Βραζιλία, το Εκουαδόρ, η Παραγουάη και αργότερα το Μεξικό ανάλαβαν τις πρώτες πρωτοβουλίες για αυτές τις συζητήσεις και Στη συνέχεια ανεπλάκησαν ε, ε, στη συζήτηση άλλες χώρες, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε λοιπόν μακρές συζητήσεις που πια ανήκουν όμως στην ιστορία Στη συγκεκριμένη φάση συζητήθηκε και το κατά πόσο χρειαζόταν μια συνθήκη και φυσικά όσοι παρακολουθήσατε τις διαπραγματεύσεις θα θυμάστε ότι αρχικά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ε, αρνητική, δεν ήθελε να υπάρξει συνθήκη. Εξελίχθηκε όμως η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την μακρά διαπραγματευτική διαδικασία όπου καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες ώστε να καταλάβουν όλοι όσοι συμμετείχαν τις προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και το 2011-12 πιστεύω ότι πια είχαμε όλοι την αίσθηση ότι προχωρούσαμε προς μια διπλωματική συνδιάσκεψη. Το Νοέμβριο του 2012 υπήρξε η βασική πρόταση, δηλαδή το κείμενο το οποίο απασχόλησε τη διπλωματική διάσκεψη και το οποίο έγιναν οι διαπραγματεύσεις. Μετά λήφθη η απόφαση για τη σύγκληση της διπλωματικής συνδιάσκεψης που ε, ξεκίνησε στο Μαρακές τον Ιούνιο του 2013. Φτάσαμε λοιπόν στο Μαρακές με ένα κείμενο που όπως πάντοτε Υπήρχαν, υπήρχε ένα ολοκληρωμένο κείμενο, κάποια κομμάτια του κειμένου εντός ε, αγγυλών και κάποια άλλα κομμάτια του κειμένου περιλάμβαναν διάφορες επιλογές. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η διπλωματική ε, συνδιάσκεψη, το επίπεδο συνεργασίας και εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις όλων των μερών ήταν ε, αξιοσημείωτο. Και μπορώ αυτό να το πω με μεγάλη βεβαιότητα γιατί συμμετείχα σε διάφορες ε, ε, διπλωματικές συνδιασκέψεις στη ζωή μου. Κάποια στιγμή λοιπόν υπήρξε κατάλληλη έφορο έδαφος και σε μεγάλο βαθμό, όπως είπα, στους οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν τους ανθρώπους αυτούς και ήταν σαφές ότι δεν μπορούσαμε να φύγουμε από το Μαρακές χωρίς να έχουμε καταλήξει σε μια συνθήκη. Και έτσι και έγινε. Η συνθήκη αντικατοπτρίζει μια συμβιβαστική λύση μεταξύ διαφόρων χωρών, διαφορετικών απόψεων, είτε αυτές ήταν απόψεις της Ένωσης, των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, του Καναδά, είτε ήταν απόψεις των Λατινοαμερικανικών χωρών, της Αφρικανικής ομάδας ή των Ασιατικών χωρών. Πιστεύω πως το τελικό κείμενο της συνθήκης είναι μια ισορροπημένη συμβιβαστική λύση Κάποιες φορές η σύνταξη θα μπορούσε να είναι σαφέστερη, αλλά ξέρετε πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις ε, στο πλαίσιο μιας διπλωματικής συνδιάσκεψης, αλλά τελικά νομίζω πως το αποτέλεσμα είναι κάτι το τελείως νέο, γιατί για πρώτη φορά α, κάναμε μια συνθήκη που ασχολείται με έναν περιορισμό, μια, μια εξαίρεση των πνευματικών δικαιωμάτων και σχετικών δικαιωμάτων, που εξασφαλίζει τη δυνατότητα διασυνοριακών ανταλλαγών. Γιατί είναι αυτό σημαντικό λοιπόν και γιατί είναι έτσι ιδιαίτερη η συνθήκη του Μαρακές. Η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε ότι χρειαζόταν αυτή η συνθήκη γιατί έπρεπε να αντιμετωπιστεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που σχετίζεται με το γεγονός ότι η κατασκευή ειδικών ε, μορφοτύπων έργων, έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση για τους ανθρώπους που έχουν ε, δυσκολία στην πρόσβαση στον γραπτό, στα γραπτά έργα, είναι εξαιρετικά δαπανηρή. Και τα μέσα που έχουν στη θέση τους όσοι εργάζονται με τους ε, τυφλούς είναι περιορισμένα. Γι' αυτό και υπάρχει ανάγκη για συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες χώρες, ανάμεσα στην Ευρώπη και όσους προσπαθούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους με οπτικές δυσκολίες σε άλλα μέρη, γιατί στην, Ευρώπη έχουμε τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά, τα ισπανικά, που μιλούνται ευρέως σε άλλα μέρη του κόσμου. Και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί το κόστος και οι δυσκολίες του να υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα και πολλά, πολλά αριθμα αντίγραφα τέτοιων έργων και να μπορούμε να εγγυηθούμε λοιπόν ταυτόχρονη πρόσβαση στον ίδιο βαθμό για τους ανθρώπους χωρίς αναπηρία και για αυτούς με αναπηρία. Γίνεται τώρα προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να κυρωθεί και να εφαρμοστεί η συνθήκη και έχουμε εμείς δραστηριοποιηθεί στην Επιτροπή για την κύρωση είναι επιτάπητος στο Συμβούλιο το θέμα Περιμένουμε την τελική συζήτηση μόλις θα γνωρίζουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το κατά πόσο είναι αποκλειστική ή κοινή αρμοδιότητας, μεικτής αρμοδιότητας μάλλον αυτή η συνθήκη και περιμένουμε την επικύρωση και από το Κοινοβούλιο σας και αυτό συζητάτε εδώ υπό τη μορφή της οδηγίας και του κανονισμού. Η Επιτροπή πιστεύει πως είναι ένα σπάκελος που πρέπει να διεκπαιρεωθεί γρήγορα και γι' αυτό και είμαστε γνώμονες για τις προσπάθειες του εισηγητή και του Κοινοβουλίου. Και αυτό επηρεάζει, πιστεύω, και το Συμβούλιο, γιατί μπορείτε να δείτε ότι καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες και από πλευρά του για να εξεταστεί αυτό το θέμα. Πριν με χτυπήσετε με το σφυράκι σας, κύριε Πρόεδρε, σταματώ. Αυτά και ευχαριστώ. Thank you. That Καλά κάνατε, λέει ο πρόεδρος. Ο πρώτος από τους κύριους προσκεκλημένους μας ομιλητές, ο κύριος Άγγερμαν. για το πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα βασικά εμπόδια της εφαρμογής στην Ένωση. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Σάγκερμαν. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας γιατί μου δίνει την ευκαιρία να μεταφέρουμε τις απόψεις μας. Κυρίες και κύριοι, εκτιμούμε δεόντως εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με δύο συγκεκριμένες προτάσεις να δώσει περισσότερες εγγυήσεις για την στρατηγική της εφαρμογής της συνθήκης του Μαρακές. Ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συμφωνήσουν μεταξύ τους το ταχύτερο δυνατόν έτσι ώστε οι προτάσεις αυτές να γίνουν δεκτές. Σχετικά όμως με κάποιες από τις προτάσεις και κάποιες τροπολογίες, η Ένωση Τυφλών έχει να μεταφέρει πολλές ανησυχίες και είναι υποχρεωμένη να απορρίψει κάποιες προτάσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο να τροποποιήσουν το σημείο 11 της προτινόμενης οδηγίας η οποία δεν σέβεται το δικαίωμα της πρόσβασης στον πολιτισμό των ανθρώπων με προβλήματα όρασης και που θα εξασθενήσει πολύ σοβαρά την πρόταση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, λεπτομερέστερα σχετικά με την εμπορική διαθεσιμότητα. Αν μπορείτε να αγοράσετε ένα αγαθό μπορείτε και να το δανειστείτε. Από ό,τι φαίνεται αυτό όμως είναι αποκλειστικότητα ορισμένων <clears throat> πνευματικών εμπλεκομένων εταίρων ε, στα πλαίσια και των συνθήκων ε, που προβλέπει η ίδια η συνθήκη του Μαρακές. Προβλέπεται να υπάρχουν μέτρα για αυτούς οι οποίοι λόγω της αναπηρίας τους δεν μπορούν να διαβάσουν τα κανονικά βιβλία. Οι βιβλιοθήκες για τους τυφλούς και τους δυσλεξικούς είναι μια βασική πηγή, θα έλεγα, προσβάσιμων βιβλίων, είτε σε προφορική εκτέλεση είτε με διαφορετικές πλατφόρμες ανάγνωσης. Κάποια κρατημέλη φαίνεται ότι είναι έτοιμα όμως να αδειάσουν τα ράφια αυτών των βιβλιοθήκων και να πούμε ότι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί να αγοράζονται εμπορικά μπορεί να ε, βρίσκονται σε αυτές τις βιβλιοθήκες. Φανταστείτε ε, πώς θα φαινόταν μια βιβλιοθήκη κανονική η οποία δεν θα μπορούσε να περιλαμβάνει βιβλία τα οποία το κοινό με τη σειρά του δεν θα μπορούσε να αγοράσει. Νομίζω ότι οι εμπορικές, αν θέλετε, εμπορικά συμφέροντα δεν πρέπει να ανατρέψουν τη συνθήκη, γιατί αυτό θα είναι φυσικά μια διάκριση εις βάρος των τυφλών. Οι πολίτες μπορούν να αγοράσουν ή να νοικιάσουν ή με ελάχιστο κόστος να, ε, εν να συμβουλευτούν ένα βιβλίο από τις δημόσιες ε, βιβλιοθήκες. Οι τυφλοί δεν θα μπορούν. Θα είναι επίσης για τις βιβλιοθήκες ένα τρομακτικό γραφειοκρατικό βάρος και θα δημιουργηθεί μια νομική αβεβαιότηση η οποία με τη σειρά της θα έλεγα απαγορεύσει την, το να συμβουλεύεται κανείς τέτοιου είδους εκδόσεις. Και δεν θα υπάρξουν και κίνητρα για τη βιομηχανία την εκδοτική διότι το Μαρακές υπάρχει λόγω ακριβώς αυτού του κενού του εμπορικού, στο οποίο η βιομηχανία δεν μπόρεσε να παράγει αυτά τα οποία απαιτούνται. Και τέταρτον, δεν υπάρχει ορισμός της λεγόμενης εμπορικής διαθεσιμότητας. Πού, με ποια τιμή και κάτω από ποια μορφή. Συνεπώς λοιπόν ουσιαστικά περιορίζεται η πρόσβαση στην πλειοψηφία των τυφλών που έχουν και περιορισμένα εισοδήματα. Δεύτερον, η λεγόμενη αντισταθμιστική αμοιβή. Ιδανικά οι εκδότες όλο και περισσότερο θα δημοσιεύουν τους τίτλους τους σε προσβάσιμα φόρματ, έτσι ώστε αυτοί που έχουν προβλήματα όρασης και άλλα προβλήματα αναπηρίας να μπορούν να τα αγοράζουν ή να τα δανείζονται από μια βιβλιοθήκη δανειστική. Όταν ειδικά όμως μιλάμε για την λογοτεχνία, για εκπαιδευτικούς λόγους ή επαγγελματικούς λόγους, εκεί δεν έχει υπάρξει κανένα βήμα προς τα εμπρός. Κάποια αυστηρά τεχνικά μέτρα δεν λύνουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι τυφλοί, με πάρα πολλά περίπλοκα, περίπλοκους πίνακες ταχύτητα περάσματος των εικόνων κτλ. Στην ουσία λοιπόν έχουμε να μιλήσουμε για μια έλλειψη πραγματικά, ένα λοιμό εκδιδόμενου υλικού. Και ξέρουμε τι έγινε και σε δίκτυα στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλους παρόχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παρέχουν, παρέχουν σειρά βιβλίων με κόστος το οποίο αναλαμβάνουν. Χρηματοδοτούνται από ιδιωτικές δωρεές και σε ορισμένες περιπτώσεις από, θα έλεγα, μικρά σχετικά δάνεια που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της κάθε χώρας. Χρησιμεύουν ε, για μη εμπορικούς στόχους, και οι οργανώσεις αυτές στην ουσία είναι οι αδειοδοτημένες αρχές οι οποίες παρέχουν στους τελικούς χρήστες το δικαίωμα ανάγνωσης όπως το προβλέπει η συνθήκη του Μαρακές. Συνεπώς κάθε απόπειρα η οποία θα είχε σαν στόχο το να περιοριστούν τέτοιου είδους δυνατότητες δεν είναι καλοδεχούμενη και ταυτόχρονα εμείς ε, ε, εκφράζουμε και λέμε ότι κάθε ή αδίποτε τέτοια προτινόμενη μορφή αντισταθμιστικής αμοιβή θα ήταν, αν θέλετε, μια επικαλυπτόμενη ουσιαστικά δαπάνη, γιατί θα έπρεπε οι επιχειρήσεις αυτές και οι οργανισμοί αυτοί να πληρώνουν δύο φορές ουσιαστικά το κόστος του έργου το οποίο παρέχουν. Το άρθρο 21 της Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αναπήρων λέγουν ότι οι προσβάσιμες πληροφορίες είναι προσβάσιμες χωρίς επιπλέον κόστος. Συνεπώς λοιπόν η αδίποτε τιμολόγιο, η αδίποτε τιμολόγηση μάλλον, ή τίμημα γενικότερα, το οποίο θα έλεγα οδηγεί σε μία επιβάρυνση της τιμής, για να καλυφθεί δήθεν το υψηλό κόστος παραγωγής θα παραβιάζει το άρθρο 21 της Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών για τους Αναπήρους. Εάν αποδεχθούμε ότι θα πρέπει οι εκδότες να είναι αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη για την διαθεσιμότητα των προϊόντων τους, τότε πραγματικά δεν υπάρχει καθόλου χώρος ε, για να διατεθούν τα προϊόντα αυτά παρά η κανονική πρώτη τιμή στην αγορά. Συνεπώς λοιπόν εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι να υπάρξει σεβασμός των κεντρικών στοιχείων της ε, προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κανονισμού τον οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πλήρη στήριση των νομικών ρυθμίσεων τις οποίες προβλέπει η συνθήκη του Μαρακές για να αντιμετωπιστεί επιτέλους η έλλειψη βιβλίων, θα έλεγα ο λοιμός των βιβλίων για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Thank you very much. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Άγγερμαν για την παρουσίαση του θέματος. Το λόγο θα λάβει τώρα θα λάβουν μάλλον οι εκπρόσωποι των εκδοτών. Ο κύριος Ζωζέ Μποργκίνο, Γενικός Γραμματεύς της Διεθνούς Ενώσεως Εκδοτών και ο κύριος Πιέρο Ατανάσιο της Ιταλικής Ενώσεως Εκδοτών, ε, Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων. Προβλέπονται 8 λεπτά και για τους δυο σας. Όποιος ε, εκ των δύο σας επιθυμεί πρώτος να λάβει το λόγο. Πρώτα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέγομαι Χωσέ Μποργκίνο, είμαι Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ενώσεως Εκδοτών και είναι η πρώτη φορά που εμφανίζομαι ενώπιον της Επιτροπής σας. Δίπλα μου είναι ο Πιέρο Ατανάσιο, τον Διευθυντής Ευρωπαϊκών Διεθνών Υποθέσεων της ε, Ιταλικής ε, Ενώσεως Εκδοτών και μέλος βέβαια της Επιτροπής μας. Ο δε κύριος Λαβιτσάρη που είναι νομικός σύμβουλος και έχει επίσης προσκληθεί να ομιλήσει δηλώνει ότι κολλείεται διότι υπερίπταται του Ατλαντικού αυτή τη στιγμή. Σύντομη εισαγωγή. Ιδρυθήκαμε το 1996 στο Παρίσι, μεγαλύτερη ομοσπονδία εκδοτών στη, στον κόσμο. Έχουμε 70 μέλη σε 60 χώρες και ε, εκπροσωπούμε χιλιάδες εκδοτών ανά τον κόσμο. Ρόλος μας είναι να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των εκδοτών, τα διάφορα copyright και υποστηρίζουμε βεβαίως την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εκδοτών. Έχουμε ήδη διαβιβάσει ορισμένα έγγραφα, τον οδηγό του Μαρακές, καθώς και την κοινή δήλωση σε αγγλικά και ιταλικά και, την, και το έγγραφο θέσεών μας για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Μαρακές. Μας προσκαλέσατε σήμερα εδώ για να απαντήσουμε αν έχουμε ξεπεράσει τα βασικά εμπόδια για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Μαρακές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύντομη απάντηση είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμβάλλει για να αποκατασταθεί μεγαλύτερη δυνατή εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών ώστε να υπάρξει πραγματική συνεργασία. Η RPA η ε, Ένωσή μας δηλαδή, από την αρχή συμμετέχει στην εφαρμογή, ήδη από τις αρχές του, του, της δεκαετίας του 2000. Είμαστε και ιδρυτικό μέλος της ABC, που είναι ένα κονσόρτσιουμ μια κοινοπραξία δηλαδή εκδοτών και θέλουμε να αυξήσουμε την ε, πρόσβαση σε βιβλία διαφόρων ε, μορφοτύπων και να ωφεληθούν βεβαίω και άνθρωποι οι οποίοι είτε τυφλοί είναι είτε έχουν μειωμένη όραση. Το 2013 ήμουν στο Μαρακές και εκεί εορτάσαμε, ε, μάλλον ε, ναι, ε, είχαμε την επέτειο της νέας αυτής ε, συμφωνίας. Έκτοτε έχουμε ζητήσει από τα μέλη μας, έχουμε συστήσει τα μέλη μας να συνεργάζονται με τις ενδιαφερόμενες αρχές. Έχουμε συστήσει από όλους τους εκδότες μας να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε εκδόσεις βιβλίων που να είναι και για τυφλούς ή μειωμένης οράσεως πρόσωπα. θέλ, επιζητούμε να διαμορφώσουμε μια διαδικασία όπου οι εγκεκριμένες αρχές σε κάθε χώρα μέλος να είναι καταχωρισμένες και να μπορούν να υπάρχει πρόσβαση σε αυτές καθώς και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό θα επιτρέψει την νόμιμη πρόσβαση, αλλά θα ρυθμίσει επίσης και θα καταστήσει διαφανή την ταχεία εργασία των εγκεκριμένων ε, ε, οντοτήτων στις διάφορες ε, χώρες και θα αποκαταστήσει το, την εμπιστοσύνη μεταξύ αυτών και των εκδοτών για να μπορούν ε, να εμφανίζονται μέσα από ένα μητρό οι εγκεκριμένε οντότητε. Αν γίνει αυτό δηλαδή θα υπάρξει καλύτερη, με καλύτερη δυνατή διακίνηση αντιτύπων, υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, θα επιτρέψει και την ανταλλαγή φακέλων με τρίτους, με διάφορες μορφές είτε και με διμερείς συμφωνίες μεταξύ των εγκεκριμένων οντοτήτων και των αναγνωρισμένων συνομιλητών τους σε τρίτες χώρες έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να παίξει έναν πρωτοποριακό ρόλο στην παγκόσμια εφαρμογή της συμφωνίας. Να μου επιτρέψετε τώρα να παραδώσω το μικρόφωνο στον συνάδελφό μου Πιέρο Ατανάσιο. Ευχαριστώ και εγώ. Εμείς ε, και από ενθουσιασμό ε, διαπνεόμαστε, αλλά έχουμε και απογοήτευση, διότι στην Ιταλία έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια. Υποστηρίζουμε τους εκδότες εμείς της Libri Italiani Accessibili, δηλαδή των, ε, προσβάσιμων μάλλον ιταλικών βιβλίων, ελέγχουμε και κάθε φάκελο που παράγουν οι εκδότες για να μπορέσουμε να, να τον αδειοδοτήσουμε ως πλήρως προσβάσιμο. Διανέμονται από τους συνήθεις διάβλους διανομής στην Ιταλία που όλοι τους γνωρίζουν και αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα για κάθε ένα από τους φακέλους. ώστε όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην, στις ίδιες πληροφορίες που μπορούμε να έχουμε όλοι μέσω οποιοδήποτε ε, παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή να μπορούν να πάνε στη βιβλιοθήκη διότι είμαστε διασυνδεδεμένοι και με το σύστημα βιβλιοθηκών της χώρας, της Ιταλίας πάντα. Αυτό έχει προξενήσει μεγάλο ενθουσιασμό σε όλους μας. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι και εκδότες και λιανέμποροι και όσοι ε, λειτουργούν τις διάφορες ε, πλατφόρμες, βιβλιοθήκες κλπ. Και ιδίω βεβαίω η Ιταλική Ένωση Τυφλών. Το αποτέλεσμα είναι ότι 40% των, δύο, των νέων μάλλον τίτλων ε, παράγονται στην Ιταλία με μορφή προσβάσιμη και σε τυφλούς και μειωμένης οράσος ανθρώπους λαμβάνουμε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία από πολλούς που μας λένε ότι αλλάξαμε τη ζωή τους. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ε, πόσο ε, μεγάλη αισθηματική, συναισθηματική μάλλον ικανοποίηση μας προκαλεί. Είμαστε πραγματικά τόσο ικανοποιημένοι που το κάνουμε αυτό. Όμως, το δεύτερο που έλεγα πριν είναι και η συνειδητοποίηση, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι 40% δεν αρκεί. Άρα χρειάζεται να βελτιωθεί το ποσοστό αυτό. Το δεύτερο είναι ότι, και συμφωνώ απολύτως με τον συνάδελφο της EBU όταν λέει ότι δεν είναι αρκετό διότι παραμένουν ακόμα πολλές ανάγκες. Υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις ακόμη. Και βεβαίως είναι αναγκαίο, αναγκαία η συνεργασία. Η εμπειρία της ενώσεως εκδοτών μας δείχνει ότι 90% των βιβλίων που εκδίδονται και που αγοράζονται για τους τυφλούς ξεκινούν από ένα master file που δίνουν οι εκδότες. Άρα μπορεί να υπάρξει και μεγάλη εξοικονόμηση και κόστους μέχρι 80%. Άρα χρειάζεται συνεργασία. Συνεργασία, ε, ανάγκη να συνομιλούμε με όλες τις πλευρές και να ακούμε και να μαθαίνουμε ημένα από τους δε. Αυτή η μακρά εμπειρία συνεργασίας μας έχει επιτρέψει να κάνουμε και μια κοινή δήλωση για τη Συμφωνία Μαρακές μεταξύ των εκδοτών, της ενός εκδοτών και της ενός τυφλών που την έχετε τη δήλωση αυτή στα αγγλικά. Γιατί ήταν εύκολο για μας και τα δύο μέρη δηλαδή να κατανοήσουμε με τους δε και να αναγνωρίσουμε για παράδειγμα ότι είναι δύσκολο να ελεγχθεί εάν προσβάσιμα αντίγραφα είναι διαθέσιμα χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύνουμε υπερβολικά τις ε, αρμόδιες οργανώσεις. Από την άλλη μεριά είναι ανόητο να κάνουμε προσβάσιμο ένα βιβλίο το οποίο είναι ήδη προσβάσιμο. Και οι δύο πλευρές όμως αναγνωρίζουμε ότι ίσως υπάρχουν περιπτώσεις όπου η συνεργασία και μπορεί να υπάρχουν ειδικέ ανάγκες διότι ένα βιβλίο που είναι προσβάσιμο σε ορισμένους δεν είναι προσβάσιμο για άλλους. Και εκεί χρειάζεται λοιπόν να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των χρηστών. Και αυτό αποτελεί θεμέλιο λίθο της συνεργασίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος κ. Ατανάσιο. Το μικρόφωνο θα λάβει ο κύριος Στίβεν Βάινμπεργκ, υπεύθυνο έρευνας των, ε, της Διεθνούς Ενώσεως Βιβλιοθηκών, πάλι για 8 λεπτά. Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω εδώ σήμερα. Εγώ εργάζομαι για τη Διεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων. Η βιβλιοθήκες κάνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά όπως μπορείτε να δείτε στις σχετικές νομοθεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στο Βέλγιο, οι βιβλιοθήκες έχουν την εντολή να εξυπηρετούν ολόκληρη την κοινότητα, πράγμα που περιλαμβάνει φυσικά και τους ανθρώπους με αναπηρίες. Υπάρχει νομικός η εντολή αυτή. Επίσης αναφέρθη ότι υπάρχουν ε, ε, βιβλιοθήκες που ειδικεύονται για τα άτομα με αναπηρίες και έχουν μεγάλο ρόλο να παίξουν γιατί ε, ας πούμε, ε, πρέπει να τηρούν κάποια πρότυπα. Επίσης συμμετέχουν στην WIPO και προωθούν για διεθνή πλαίσια για τα πνευματικά δικαιώματα για καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες των χρηστών και τις ανάγκες των εκδοτών, ώστε να υπάρχει και οικονομική ευημερία. Ο στόχος μας εδώ είναι μια κατάσταση όπου ο Λοιμό των βιβλίων να ανήκει στο παρελθόν. Έχουμε πολλά καλά παραδείγματα, τα όσα γίνονται στην Ιταλία και το έχω ακούσει και από άλλε πηγέ, μπορώ δηλαδή να το επιβεβαιώσω ότι όντω συμβαίνει αυτό. Η Ιταλία είναι ένα καλό παράδειγμα. Πάει καλά το πράγμα, αλλά φυσικά δεν συμβαίνει παντού. Περνάμε από μια κατάσταση από πλήρου αποτυχία τη αγορά, που είναι απαραίτητο για να βγούμε από αυτή την κατάσταση και να προωθήσουμε την πρόσβαση με οποιονδήποτε τρόπο είναι κάτι το θετικό. Έχουμε τέσσερις-πέντε συστάσεις. Ε, πρώτον, να εστιαστούν οι πόροι. Όπω είπε ο κύριο Άγγερμαν, οι βιβλιοθήκες είναι οργανισμοί που εργάζονται με περιορισμένου δημόσιου προπολογισμού. Ε, οι οργανισμοί που τυπώνουν για τους ανθρώπους με δυσκολίες όρασης επίσης λειτουργούν με περιορισμένο προπολογισμό. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό κάθε ευρώ να δαπανάτε με αποτελεσματικό τρόπο ώστε να υποστηριχθεί πρόσβαση. Δεν λέμε ένα για τσάμπα δωρεάν πράγματα, όχι. Οι βιβλιοθήκες πληρώνουν για το περιεχόμενο που έχουν, αλλά και το ίδιο και οι ειδικοί οργανισμοί. Όταν πρέπει να φτιάξουν ένα ειδικό μορφότυπο όμω, το κόστο ανεβαίνει σε χιλιάδε ευρώ. Γι' αυτό όταν έχουν και το αντίτυπο και την προσβάσιμη μορφή του, εάν μετά χρεώνουμε για την πρόσβαση, αυτό μειώνει τη δυνατότητα των, ε, θεσμο, των ιδρυμάτων αυτών να κάνουν ό,τι μπορούν το καλύτερο για τους χρήστες τους. Έπειτα θα πρέπει να προσφερθεί μια βεβαιότητα στα ε, ιδρύματα αυτά. Ε, ε, αυτό σε σχέση με τους ελέγχους εμπορικής διαθεσιμότητας περιλαμβάνεται στο ε, άρθρο 11. Στην ουσία αυτό το ερώτημα είναι κάτι το κενό γιατί όταν έχεις μια βιβλιοθήκη, έναν εκδότη μάλλον που είναι έτοιμος να προσφέρει το αντίτυπο και να προσφέρει και το ειδικό μορφότυπο, ε, τότε δεν έχει νόημα. Η εμπειρία από την Αυστραλία που έχουμε δείχνει ότι αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για την εμπορική διαθεσιμότητα, ε, Ξεκάθαρο ορισμός, αυτό μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο. Γιατί στην Αυστραλία, α πούμε, ε, τι έγινε, αν έχουμε την απέτηση εμπορική διαθεσιμότητα, αυτό σε αναγκάζει να ε, πολύ πολυάριθμα αντίτυπα πρόσβαση. Όμω το αντίγραφο δεν είναι στο καλό μέγεθο, δεν είναι αρκετά μεγάλο για τον χρήστη, πάλι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξαίρεση. Ακόμα και αν το διαθέσιμο αντίτυπο δεν είναι αρκετά καλό. Και το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό εάν κανεί σκεφτεί τι διασυνοριακέ ανταλλαγέ. Βλέπουμε ότι το να βρει κανεί αν υπάρχει εμπορικά διαθέσιμο σε μια, ένα βιβλίο σε μια αναπτυσσόμενη χώρα είναι αδύνατον σχεδόν αν θέλουμε να μπορέσουν συγκεκριμένες μονάδες στην Ευρώπη να υλοποιήσουν το δυναμικό τι συνθήκε του Μαρακέ διεθνώ. Δεν μπορούμε να του αναγκάζουμε να περνούν από αυτή τη διαδικασία κάθε φορά δηλαδή να αναζητούν ε, τα διαθέσιμα τίτυπα. Επίση είναι θέμα εγκύτητα στου χρήστε και επανερχόμαστε στο θέμα των δημοσίων βιβλιοθηκών που έχουν υποχρεώσει να εξυπηρετούν ολόκληρη την κοινότητα στην οποία βρίσκονται. Να γνωρίζουν του χρήστε και να παρέχουν τι απαραίτητε υπηρεσίε. Είναι μια βασική αρχή τη ε, Σύμβαση για τη Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρίε. Οι ίδιε υπηρεσίε θα έπρεπε να υπάρχουν για όλου προσαρμόζονται σε όλους. Οπότε οι δημόσιες βιβλιοθήκες, η βιβλιοθήκη της γωνιά, θα πρέπει, ε, στο δρόμο θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει αυτές τι δυνατότητες. Στη στιγμή που κανείς μπορεί, να πάει να ψάξει και να γραφτεί στην βιβλιοθήκη θα πρέπει να έχει τη στη διάθεσή του τα βιβλία. Και το άρθρο 9 τη συνθήκη λέει σαφώ ότι αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτική εγγραφή δεν υπάρχει εκεί και δεν προβλέπεται και δεν πρέπει και να το κάνουμε γιατί αυτό θα φοβήσει τον κόσμο ακόμα και αυτόν που είναι έτοιμος να βοηθήσει τους ανθρώπους με αναπηρίες. Και μιλήσαμε για εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι για τις βιβλιοθήκες είναι ενδιαφέρον αυτό το θέμα γιατί μιλάμε για ένα δίκτυο επαγγελματικών οργανώσεων που στελεχώνονται από ειδικευμένους ανθρώπους και δεσμεύονται από επαγγελματικούς κώδικες διοντολογία. Αν δείτε τα όσα λέει η συνθήκη, αυτό κάνουν ούτω ή άλλω ήδη οι βιβλιοθήκε. Δηλαδή να εξασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τα βιβλία ε, είναι επιλέξιμοι. Έχουν τι κάρτε τη βιβλιοθήκη, του ενθαρρύνει και βρίσκει τρόπου να, να σταματήσουν οι παραβάσει. Και αυτό το κάνουν καθημερινά οι βιβλιοθήκε. Εξασφαλίζει ότι έχει ε, μητρό ε, και πάλι οι βιβλιοθήκες ήδη το κάνουν αυτό και συμφωνία με το όσο έλεγε νωρίτερα ο κ. Σάγκερμαν, εάν επιβάλλουμε επιπλέον υποχρεώσεις και απαιτήσει στις βιβλιοθήκες θα καταστεί πιο δύσκολη η δουλειά τους. Και αυτό αναφέρεται πάλι και στη σύμβαση για τους ε, ανθρώπους με αναπηρία. Ξέρουμε ότι γίνεται πειρατεία στον κόσμο, αυτό υπάρχει. Όμως να σας πω από ένα σεμινάριο που έγινε στη Γουάιπο πέρυσι ότι οι επικεφαλής αρμόδιοι για τη διανομή και για την προσβασιμότητα αντιτύπων ε, βιβλίων στην Ινδία, στην Αργεντινή, στη ΣΥΠΑ, όταν τους ρωτήθηκε αν υπάρχουν αποδείξεις για συστηματική και μεγάλη πειρατεία, όλοι απάντησαν όχι. Δεν είναι κάτι το οποίο σημαίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τέλος, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη δίνουν ε, το παράδειγμα στον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρώπη ε, ε, δίνει το παράδειγμα και ο υπόλοιπος κόσμος στην ουσία αντιγράφει αυτά που κάνει η Ευρώπη. Επιπλέον αμοιβή η εμπορική διαθεσιμότητα λοιπά, Αν είναι δύσκολα στην Ευρώπη, αλλά για μια βιβλιοθήκη, για μια βιβλιοθήκη σε μια ανεψόμενη χώρα, αυτό θα, το, θα την διαλύσει τελείω. Ε, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Θα πρέπει να θυμόμαστε λοιπόν, όταν εδώ περνάμε νομοθεσία, ότι ό,τι κάνουμε έχει αντίκτυπο στον υπόλοιπο κόσμο θα πρέπει να φροντίσουμε ό,τι κάνει η Ευρώπη να μην επηρεάσει αρνητικά το δυναμικό της συνθήκης του Μαρικές. Και πιστεύω ότι είναι σπάνιο από έναν Βρετανό, οι συνάδελφοι στην Κομισιόν είπαν ότι είναι σπάνιο ε, να πούμε ότι η δουλειά που έκανε η Κομισιόν ε, αρχικά ήταν πολύ καλή δουλειά. Θέλουμε κάποια μικροπράγματα να αλλάξουν, αλλά ξεκινάμε από πολύ καλό σημείο θετηρία. Και προ χάρη τη γρήγορη κύρωσης αυτού του κειμένου, α μείνουμε σε αυτό, α μην το αλλάξουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. And Ήρθε η ώρα να μπορέσουν να θέσουν τα μέλη ερωτήσεις, αν επιθυμούν. Δεν βλέπω κανένα. Θα ρωτήσω εγώ τότε. Μπορείτε να μας υπενθυμίσετε πόσοι δυνατοί δικαιούχοι, πόσοι πιθανοί δικαιούχοι υπάρχουν. Δηλαδή πόσα πρόσωπα μπορεί να υποφεληθούν από την εφαρμογή της Συμφωνίας του Μαρακές. Έχετε νούμερα. Με επιτρέπετε ο κύριος Άγγερμαν. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σύμφωνα με υπολογισμούς υπάρχουν 285 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο που είναι είτε τυφλοί είτε μειωμένοι οράσος. Στην ΔΕ Ευρώπη ο αριθμός αυτός υπολογίζεται σε 30 περίπου εκατομμύρια ανθρώπους ανά την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη. Με όλων των βαθμών μερική όραση, όπως ε, ε, τους χαρακτηρίζουμε στην Ευρώπη. Βέβαια και υπάρχει και αριθμός απολύτως τυφλών ανθρώπων, οι οποίοι όμως είναι πολύ μικρότεροι, ε, πολύ μικρότερος αριθμός από αυτά τα 30 εκατομμύρια. Είναι δύσκολο να δοθούν ακριβή νούμερα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρέντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ επικοδομητική η παρουσίασή σας. Αφού άκουσα προσεκτικά, η πρώτη αίσθηση που μου δημιουργήθηκε είναι ότι υπάρχει αρκετή σύγκληση ανάμεσα στις διαφορετικές θέσεις. Μία ερώτηση προς τον κύριο Άγγελμαν. Αναφερθήκατε στην Ομοσπονδία των Ευρωπαίων Εκδοτών, οι οποίοι μας μετέφεραν και τις απόψεις τους, ε, θεωρούν ότι το 11 θα πρέπει να αναθεωρηθεί και ότι μόνο τα εμπορικά διαθέσιμα έργα θα είναι προσβάσιμα σύμφωνα με τη συνθήκη του Μαρακέσου. Τώρα, οι βιβλιοθήκες ε, ειδικά για ανθρώπους με προβλήματα όρασης, θα διαθέτουν φυσικά και εμπορικά προϊόντα, αλλά το θέμα είναι ποιος είναι ο νόμος που εφαρμόζεται σε κάθε χώρα. Κάτι το οποίο είναι δημόσια προσβάσιμο σε μία χώρα δεν είναι σε μία άλλη. Οπότε πώς είναι δυνατόν ε, οι βιβλιοθήκες και οι διάφορες οργανώσεις στην κοινωνία των πολιτών ε, τι μέτρα μπορούν να πάρουν για να γνωρίζουν ακριβώς τι δυνατότητες έχουν και τι είναι εφικτό ουσιαστικά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, λέει ο κύριος Σάγκερμαν. Όταν έχετε κάποιες συγκεκριμένες αποδείξεις ότι έχει δημοσιευθεί ένας τίτλος, ένα βιβλίο, γνωρίζετε ότι υπάρχει θεωρητικά εμπορική διαθεσιμότητα. Το θέμα όμως δεν είναι τόσο περίπλοκο. Ένα τυφλός, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα διαθέσιμο τίτλο, θα το κάνει αυτό. Και το βιβλίο αυτό φυσικά θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και σε συγκεκριμένες βιβλιοθήκες. Αλλά ποτέ καμία βιβλιοθήκη όταν έχει έναν τίτλο διαθέσιμο δεν θα χρησιμοποιήσει την δυνατότητα να αγοράσει τον ίδιο τίτλο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχετε ας πούμε ένα βιβλίο, ένα φάκελο ο οποίος φαίνεται ότι είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά τουλάχιστον θεωρείται ότι είναι διαθέσιμος, ενώ στην πραγματικότητα θα καταλάβετε ότι αυτά τα PDF δεν είναι πια διαθέσιμα, γιατί έχουν, ε, αν θέλετε, μια αρχιτεκτονική ανάγνωση η οποία είναι σε στήλε και η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτόν που έχει προβλήματα όρασης. Συνεπώς λοιπόν τα τεχνικά προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα πρέπει η αδειοδοτούσα αρχή να καθιστά με τα μέτρα που χρειάζονται διαθέσιμους τους τίτλους αυτούς. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Το όνομά σας παρακαλώ. Είμαι ο Ντέβιτ Χάμερστιν. Εκπροσωπώ την Διεθνή Ένωση Τυφλών. Είμαι πραγματικά ευτυχής για αυτά τα οποία άκουσα. Έχουμε φτάσει, θα έλεγα, σε μια ιστορική καμπή για τη συνθήκη του Μαρακές. Η συνθήκη του Μαρακές θα είναι χρήσιμη και θα ωφελήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, εάν επικυρωθεί και εφαρμοστεί σωστά από την Ένωση, γιατί αλλιώς δεν θα πάμε καλά. Ε, πράγματι μας επιβεβαίωσαν με επιστολές τους ε, διάφοροι ότι οι Γερμανοί εκπρόσωποι της κυβερνήσεως ε, πιέζουν για να γίνει κάτι το οποίο ο κύριος Μπαρνιέ είχε πει ότι δεν θα πρέπει να ε, συμβεί. Δηλαδή από τη μία να έχουμε τις ρήτρες τις λεγόμενες του Μαρακές και από την άλλη να έχουμε τις ρυθμίσεις για αποζημιώσεις στα πλαίσια της πνευματικής ιδιοκτησίας να υπάρξει δηλαδή μια ανάμιξη των δύο, νομίζω ότι δεν είναι η εύθετη στιγμή έτσι ώστε να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιβαρύνουμε τη συνθήκη του Μαρακές με μια προβληματική πολύ γενικότερη. Ακούγονται διάφορα από τη γερμανική κυβέρνηση και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κάπως το θέμα να μην ε, περιπλέξουμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να έχουμε προτάσεις οι οποίες πολιτικά θα προκαλέσουν διαιρέσεις. Στην φάση που βρισκόμαστε τώρα δεν συζητάμε γενικά θέματα copyright. Μιλάμε για ειδικά δικαιώματα, για μια ειδική κοινότητα πολιτών περιορισμένη η οποία έχει σαφέστατα προβλήματα πρόσβασης σε αναγνωστικό υλικό. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να πούμε στους Γερμανούς ότι δεν είναι η ώρα να τα συζητάμε αυτά. Ο κύριος Μπογκίνιο. Να σχολιάσω λίγο την έννοια της εμπορικής διαθεσιμότητας. Τώρα αν ένας εκδότη στον κόσμο ο οποίο δεν θέλει να προμηθεύσει μια συγκεκριμένη αγορά, σαν ιδέα αυτό δεν στέκει. Όλοι οι εκδότες που γνωρίζω θέλουν να δώσουν όσο περισσότερα βιβλία με οποιαδήποτε φορμά, σε οποιαδήποτε δυνατή μορφή, σε όσους περισσότερους πελάτες γίνεται. Συνεπώς λοιπόν εγώ δεν βλέπω τις βιβλιοθήκες να αδειάζουν ε, ειδικά για αυτούς που έχουν προβλήματα όρασης. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να βασιστούμε στην επαγγελματικότητα των εκπροσώπων των βιβλιοθηκών, να βρουν κάποιες λύσεις στα προβλήματα που έχουν και στα πλαίσια των διαθέσιμων εμπορικά και μη εμπορικά τίτλων από όλο τον κόσμο. Αυτά όλα με το διαδίκτυο μπορούν να τα βρουν με μεγάλη ευκολία να ξέρουν τι είναι διαθέσιμο και τι δεν είναι. Το βασικό θέμα το οποίο οι εκδότες θέλουν να τονίσουν σε σχέση με την εμπορική διαθεσιμότητα είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα κόσμο με πόρους οι οποίοι είναι χαμηλοί και χαμηλώνουν συνεχώς και δεν έχει νόημα να υπάρχουν πραγματικά απεριόριστοι αν θέλετε αριθμοί τίτλων όπως ε, οι τίτλοι που διαβάζονται κυρίως από παιδιά σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Το θέμα είναι να καλύψουμε το σύνολο των διαθεσίμων τίτλων. Λοιπόν, πριν κλείσει η συζήτηση, μία ερώτηση προς τον κύριο Βέιμπερ. Αλλά δεν ξέρω και αν οι εκπρόσωποι των εκδοτών θα ήθελα να απαντήσουν. Έτσι όπως εγώ βλέπω τα πράγματα, ένα από τα βασικά θέματα αυτών στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Βάιμπερ είναι ότι αν πραγματικά στραφούμε κατά των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε αν ένας τίτλος είναι εμπορικά διαθέσιμος, ή αν για να γίνει κάτι τέτοιο τεθούν και άλλα θέματα υποσυζήτηση όπως σαν παράδειγμα οι εναλλακτικέ ή συμπληρωματικέ μορφές αμοιβή του δικαιούχου κτλ. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόσει στο χαρτί τουλάχιστον τη συνθήκη του Μαρακές φοβάμαι ότι ε, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα αν θέλετε όθησης από πλευράς της εφαρμογής αυτής έτσι ώστε περισσότεροι τίτλοι να καταστούν διαθέσιμοι στον κόσμο αυτών που έχουν προβλήματα όρασης. Συνεπώς λοιπόν η εφαρμογή της συνθήκης του Μαρακές είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να μείνει στο χαρτί και θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Βάιμπερ ή οι εκδότες θέλουν να κάνουν κάποιο σχόλιο. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας, λέει ο κύριος Βάιμπερ. Οι εκδότες των τίτλων που θα καταστούν διαθέσιμοι, ακόμα και αν αυτή, όπως είπα, η έλλειψη, η σπάνης τίτλων είναι κάτι το οποίο φτάνει μερικές φορές σε τρομερά ποσοστά όπως το 1%. Δεν μπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις για την διαφυσιμότητα των τίτλων. Ε, τα παραδείγματα τα οποία έχουν μας δίνουν ότι υπάρχουν εθνικές ρυθμίσεις ε, οι οποίες ε, μπορεί να βρουν λύσεις, αλλά σε διεθνές επίπεδο είναι κάτι το οποίο ε, ίσως ο διεθνός να μην μπορεί να γίνει αποδεκτός. Αν παράδειγμα στην Κολομβία έχουν ένα σύστημα copy-paste, το οποίο δύσκολα θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές. Ο κύριος Ατανάσιο, έχετε δίκιο και εσείς και ο κύριος Άντερσον όταν λέτε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον κόστος για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας σημεί. Ταυτόχρονα όμως και εσείς στο δικό σας έγγραφο, κύριε Βάιμπερ, αναγνωρίζετε ότι δεν έχει νόημα το να γνωρίζει κανείς τυπικά αν είναι διαθέσιμο ένα βιβλίο και αν θα πρέπει να υπάρξει ένα αντίγραφο που θα προκαλέσει επιπλέον κόστος. Είναι πρακτικό το θέμα και θα πρέπει να βρεθεί λύση και οι εξαιρεσει δεν νομίζω ότι μπορούν να θεωρηθούν ως κανόνας. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα μέτρα που θα ληφθούν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναντίον των χρηστών, περιοδίζοντας ακόμα περισσότερο τους τίτλους τους οποίους ε, έχουν στη διάθεσή τους. Η διαθεσιμότητα της πληροφορίας και η σωστή ενημέρωση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί όχι μόνο με τις εξαιρέσεις. Και να πω ότι ευρύτερα η συζήτηση για την διαθεσιμότητα μίας πληροφορίας είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί μέσα από την πράξη για την διαθεσιμότητα τίτλων. Νομίζω ότι εδώ είναι κάποιες συστάσεις οι οποίες θα πρέπει να δοθούν. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κάνει τώρα πια κάποια σχόλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Άλλωστε, η συναρφούς Μαρία έχει κάνει μια θαυμάσια εισαγωγή. Θα ήθελα μόνο να επιβεβαιώσω ότι εν γέννη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται το θέμα Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και διαμορφώνεται η γενική συνένεση ότι χρειάζεται να ξεβρεθεί μια εύλογη λύση σύντομα και χωρίς να προκληθεί ε, περισσότερη σύγχυση και περιπλοκή. Αυτό είναι το μήνυμα και των δύο θεσμικών σας οργάνων. Ε, είμαστε δε πεπισμένοι ότι μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Γενικότερα και βεβαίως και το θέμα της αιτιολογικής ε, σκέψης 11 και της διαθεσιμότητας στην αγορά που είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητηθεί και στην νομοθετική διαδικασία. Από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορώ να προσθέσω το εξής. Ούτε θεωρούσαμε, ούτε θεωρούμε ότι λόγω της ειδικότητας, του ειδικού χαρακτήρα δηλαδή του αντικειμένου θα χρειαζόταν καν να θεσπίσουμε αυτές τις ε, απαιτήσει, διάφορε συζητήσει σχετικά με την καταλληλότητα, με την ψηφιακή ανάλυση κλπ. Ε, θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι μιλούμε για μια ειδική κατάσταση αποτυχίας της αγοράς, όπου δεν καλύπτει δηλαδή τις ανάγκες η αγορά και πρέπει να φροντίσουμε να προσφέρουμε κάλυψη σε συγκεκριμένους ανθρώπους που είναι οι ενώσεις τυφλών και σε μια αγορά που ενδεχομένω υπάρχει, το, υπάρχει ο κίνδυνο να υπάρχουν διαφορετικέ νομοθετικέ προσεγγίσεις σε διάφορες ε, χώρες μέλη. Η προσβασιμότητα θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη. Αυτό για μας είναι ειδική περίπτωση αποτυχίας της αγοράς. Και θέλουμε να κάνουμε την εφαρμογή της συνθήκης όσο το δυνατόν απλούστερη. Αυτά μπορώ να πω για το σύγχρονο θέμα και κατά τα λοιπά. Είμαστε επεπισμένοι ότι θα καταλήξουμε σε μια λογική λύση και, όχι, και δεν θα αργήσει αυτό πολύ. Ο Πρόεδρος. Ελπίζω ότι έτσι ε, απαντήσαμε ε, σιωπηρά κατά κάποιο τρόπο και στις ε, παρατηρήσεις του κ. Μπαρνιέ που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ο κ. Άντερσον, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω ολόκληρο το πάνελ για τις διαφωτιστικές του τοποθετήσει, Εμένα μου φάνηκαν, φάνηκε όλο το θέμα δηλαδή, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και επειδή μιλούμε, και θα μιλήσουμε βέβαια, για τους φακέλους που από τη συνθήκη του Μαρακές, από αύριο θα είμαι τώρα πολύ σύντομο. Θα θέλαμε όλοι νομίζω να δούμε τη συνθήκη του Μαρακέσου να αποδίδει πραγματικά, δηλαδή να καταστούν τα έργα αυτά προσβάσιμα. Πρέπει να φροντίσουμε να γίνουν σεβαστοί οι στόχοι της συνθήκης του Μαρακέσου που έχουν συζητηθεί σε ανώτατο επίπεδο από τους οργανισμούς copyright να μην αποδυναμωθούν από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διασφαλίσουμε ώστε να μην δημιουργηθούν έξτρα περιορισμοί οι οποίοι θα υπερβαίνουν το τρέχον νομικό πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για το copyright καθώς και των Ηνωμένων Εθνών που κυρίως για τα δικαιώματα ε, ε, των αναπήρων. Ευχαριστώ πολύ, αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, τους διακεκριμένους ομιλητές και επισκέπτες μας για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απόψεις που εκφράσατε και ελπίζομαι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του θέματος επιτυχώς και σύντομα, ώστε να μην χρειαστεί να ξανασυναντηθούμε κιόλας. Θα δώσω λίγα λεπτά στους επισκέπτες μας ε, για να αποφασίσουν αν θα μείνουν στην αίθουσα ή αν θα αποχωρήσουν. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμα εργασιών μας. Μπορείτε, εάν επιθυμείτε, να συνεχίσετε να συζητείτε το θέμα που μας απασχόλησε τώρα, εκτός ευθούσης. Εσείς, κύριε Άντερσον. Να συνεχίσουμε σας παρακαλώ. Uh, now we are at υπαριθμών 4 ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικανικής Εκπαιδεύσεως. Είναι κοντά μας ο κύριος Βοστσούλσκι, Γενικός Γραμματεύς του Εν Λόγω Δικτύου, η κυρία Βαλερίσα Αγκάμ, αναπληρώτρια διευθύντρια της ε, ανώτατης σχολής δικαστών στη Γαλλία και άλλα πρόσωπα. Έχετε λοιπόν στο σύνολο 20 λεπτά για τις παρουσιάσεις σας. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί σας. Θα μοιραστούμε τα 27 λεπτά με την Βαλερή. Να αρχίσω πρώτος εγώ. Η δική μας ιδέα για την παρούσα συζήτηση είναι να θέσουμε ε, ας εξηγήσουμε τι είναι το δίκτυο ε, δικανικής ε, εκπαιδεύσεως και ποιες είναι οι προκλήσεις του EJTN 15 χρόνια τώρα έχουμε την υποστήριξή σας και να ρίξουμε και στο μέλλον και της δικανικής εκπαιδεύσεως και του EJTN. Από δύο μεριές, από δύο πλευρές θέλαμε να φωτίσουμε το θέμα που φωτίζουν το τι είναι το EGATN τώρα. Και η πρώτη σκοπιά είναι, είναι η εθνική. Η συνάδελφός μου Βαλερή θα σας εξηγήσει ε, την κατάσταση από τη δική της εθνική σκοπιά, τους, ε, τους, τους ε, θεσμούς, τα εθνικά όργανα εκπαιδεύσεως κλπ. Εγώ θα αρχίσω δίνοντάς σας κάποια στοιχεία από την σκοπιά των Βρυξελών, του Γενικού Γραμματέως του EJTN, ώστε να κατανοήσουμε όλοι καλύτερα που βρισκόμαστε με την εκπαίδευση δικαστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συμφωνήσετε και συμφωνούμε όλοι ότι τα δικανικά συστήματα απασχολούν πολύ όλους και όλες στην Ευρώπη και τι αναμένει το κοινό από εμάς, δικαστές, εισαγγελίε κλπ. Οι οποίοι καλούμεθα να εκτελούμε τα καθήκοντά μα με σοφροσύνη και επαγγελματισμό. Και βεβαίω να ελεγχόμεθα κιόλα. αυτό είναι ο ρόλο του EJTN. Το EJTN είναι ένωση και βρισκόμαστε στην καρδιά των διαδικασιών αυτών, να προετοιμάζουμε δηλαδή δικαστέ και εισαγγελεί να ανταποκρίνονται σε όλε αυτέ τι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Το JTN είναι ε, οργάνωση καταχωρισμένη εδώ στο Βέλγιο. Ε, εκπαιδεύουμε δικαστέ και εισαγγελεί σε όλε τι χώρε μέλη, με όλε τι σχετικέ ενώσει να είναι μέλη μα. Και έχουμε και την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, τη TRIER, στη Γερμανία. Ο τρόπος με τον οποίο ιδρυθήκαμε και εξακολουθούμε να λειτουργούμε απηχεί την ανεξαρτησία πρώτα-πρώτα της δικαιοσύνης. Δεν είμαστε μέλη του θεσμικού πλαισίου. Είμαστε αυτό που θέλει να είμαστε η δικαιοσύνη. Το JTN με λίγα λόγια τι είναι. Εδώ θα πρέπει να τονίσω δύο βασικά χαρακτηριστικά. Αφενός ως δίκτυο είμαστε μια ισχυρή και αποτελεσματική δομή με έδρα εδώ. Παρέχουμε τις υπηρεσίες εκπαιδεύσεως 6.000 δικαστές και εισαγγελείς τον χρόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ένας πολύ ισχυρός θεσμός. Από την άλλη μεριά, αν εξετάσει το JTN, οφείλουμε να πούμε ότι εμείς είμαστε ένα δίκτυο και αυτό είναι το βασικό μας χαρακτηριστικό. Δίκτυο των εθνικών αρχών, φορέων, παροχής εκπαιδεύσεως. Και εδώ εμείς απηχούμε το τι ζητούν οι δικαστές από εμάς. Και δεν υπαγορεύει η Γενική Γραμματεία άνωθεν αυτό το πράγμα. Περιμένουμε εκ των κάτω να μας πούν τι χρειάζονται σε όλα τα δικαστήρια και των 28 χωρών μελών, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε στο σύνολό μας όσα δεν μπορεί να, κάθει να κάνει κάθε εθνικός φορέας στην χώρα του. Να αναπτύξουμε δίκτυα μεταξύ των θεσμικών οργάνων, ώστε να διευκολυνθούν οι δικαστέ και οι εισαγγελεί να εκτελέσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα καθήκοντά του. Αυτά είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του δικτύου όπω έχει εξελιχθεί, όπω είπα πριν, την τελευταία 15 ετία τη ύπαρξή του. Το δίκτυο δεν μπορεί να υπάρξει στο κενό, χρειάζεται συνέργειε με πολλού εταίρου, βεβαίω τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα του χώρου δικαιοσύνη και εσωτερικών, για παράδειγμα ΣΥΠΟΛ, ε, όπου διεξάγουμε πάρα πολλές συνεργασίες διότι οι εισαγγελείς ε, εκπαιδεύονται μαζί με τους αστυνομικούς διότι συνεργάζονται πολύ στενά. Δεν θα αναφέρω όλες τις ενώσεις και όργανα που συνεργάζονται μαζί μας, δεν θα τα αναφέρω όλα. Συνεργόμαστε όμως γιατί ποιος, ποιο είναι το βασικό, ο βασικός πυρήνας των δραστηριοτήτων μας έχουμε μεγάλο αριθμό δικαστών από όλες τις χώρες μέλη. Αυτό είναι ένα πρώτο χαρακτηριστικό. Σε κάθε εκδήλωση που διοργανώνουμε έχουμε παρούσες τουλάχιστον 20 με 22 εθνικότητες. Δικαστές οι οποίοι συνεργάζονται στην εκπαίδευση, συζητούν, αναζητούν κοινέ λύσεις στις υποθέσεις που έχουν μεταξύ των χωρών τους. Καλύπτουμε και ένα τεράστιο φάσμα θεμάτων, όχι βεβαίω μόνο νομικά θέματα, Βεβαίω και τα θέματα της νομικής συνεργασίας που μα απασχολούν διαρκώ, αλλά και τι προκλήσεις, για παράδειγμα δίκαιο ασύλου, μετανάστευση, τρομοκρατία για του χρόνου που βλέπουμε μια εικοσαριά δραστηριότητε, ώστε να μπορέσει το δίκτυο να συμβάλλει στι απαντήσει, αυτές. Δίνουμε μεγάλη σημασία και σε μη νομικά θέματα. Προπαρασκευή, για παράδειγμα, των δικαστών για να είναι πρόεδροι δικαστηριών τους παρέχουμε γλωσσική εκπαίδευση, μαθαίνουν ξένες γλώσσες, αλλά και μεθοδολογία εκπαιδεύσεως. Δηλαδή συνομιλούμε μεταξύ μας πώς να προαγάγουμε καλύτερα και με όσο το δυνατόν λιγότερο δαπανηρό τρόπο τις σχετικές εκπαιδεύσεις και επαναλαμβάνω για τις 28 χώρες Το κάνουμε για τους δικαστές, εισαγγελείς, αλλά και τους μελλοντικού δικαστές και εισαγγελείς, αλλά και τους εκπαιδευτές στα διάφορα σεμινάρια. Αυτές με λίγα λόγια είναι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητές μας. Τι προσφέρουμε. Σας έχουμε διανύμει σήμερα την έκθεση δραστηριοτήτων μας όπου θα δείτε με λεπτομέρειες όλα τα στοιχεία και όλα τα θέματα που καλύπτουμε. Πώς εξελίχθη η προσφορά μας την προηγούμενη χρονιά. Το 2005 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να αναπτυχθεί το δίκτυο. Τότε είχαμε 160 συμμετέχοντες, 160 δικαστές, τους οποίους στείλαμε για δύο εβδομάδες σε άλλη χώρα μέλους για να δουν πώς εργάζονται οι ομόλογοι τους σε άλλες ε, χώρες μέλη. Πέρσι είχαμε πάνω από 2.000 δικαστές οι οποίοι συμμετέσχουν σε αυτές τις ανταλλαγές. Βλέπετε λοιπόν πόσο πολύ διευρύνθηκε η προσφορά μας και πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη ή οι ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ανταλλαγές αυτές και διαρκώς μεγαλώνουν. Τώρα, λίγα νούμερα, ελπίζω ότι μπορείτε να τα δείτε. Θα δείτε και την αύξηση, όχι μόνο των ανθρώπων που εκπαιδεύομαι, αλλά το γράφημα αυτό δείχνει και πόσο σημαντική είναι η προσφορά του UGTN. Με κιανό χρώμα βλέπετε τον αριθμό δικαστών και εισαγγελέων που συμμετέχουν στα διάφορα χρόνια στις διαμεθοριακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Με κόκκινο χρώμα βλέπετε τους συμμετέχοντες σε διαμεθοριακές δραστηριότητες εκτός του πλαισίου EGATN. Βλέπετε λοιπόν ότι πολύ μεγάλη πλειοψηφία συμμετεχόντων σε διαμεθοριακές δραστηριότητες είναι αυτή στις οποίες απευθυνόμεθα μέσω του EJTN. Πέρσι το 2016 φτάσαμε τους 6 περίπου χιλιάδες συμμετέχοντες στις εκπαιδευτικές δραστηριότητές μας. Βεβαίω, για να τα πετύχουμε όλα αυτά, δεχόμαστε όλο και μεγαλύτερη χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτό θα έρθω στο τελευταίο μέρος της ομιλίας μου. Το EGTN συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ε, e-Justice και ο προϋπολογισμός θα φτάσει στα 10 εκατομμύρια ευρώ. 96% των χρημάτων αυτών Μα τα δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 4% είναι η συνεισφορά των εθνικών φορέων δικαστική εκπαιδεύσεω των χωρών μελών. Μιλούμε για χρήματα, αλλά τα μέλη μας μα προσφέρουν πολύ περισσότερα, διότι μας στέλνουν και εμπειρογνώμονε, οργανώνουν εκπαιδεύσει δηλαδή είναι και συνεισφορά σε είδο και όχι μόνο σε χρήματα. Όμως χωρίς την τεράστια υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα μπορούσαμε να τα προσφέρουμε όλα αυτά. Μπορούμε όμως τώρα λόγω της σηματοδότησης αυτή να προσφέρουμε και όλο και υψηλότερη ποιότητα. Ο προπολογισμό του JTN αυξάνεται. Μπορούμε όμως και μειώνουμε και το κόστος ανά ημέρα εκπαιδεύσεως, διατηρώντας υψηλή την ποιότητα. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία και αριθμοί από την ευρωπαϊκή οπτική το, της προσφοράς του ε, δικτύου. Επιτρέψτε μου να δώσω τώρα το λόγο στην Βαλερή Σαγκάν που είναι αναπληρώτια διευθύντρια της Εθνικής Σχολής Δικαστών και να σας εξηγήσει τα πράγματα από την σκοπιά του Εθνικού Φορέα. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γαλλικά. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Αντιπρόεδροι, Κυρίε και κύριοι, εγώ ήθελα να σας δώσω την εικόνα ενό από τα μέλη αυτού του δικτύου, διότι η Εθνική Σχολή Εισαγγελέων της Γαλλίας στηρίζει, είναι, κομμάτι, είναι μέλος αυτής του, αυτού του δικτύου και στηρίζει δραστηριότητε του από τη δημιουργία του. Και δόθε είναι πολύ γνωστή η συμβολή, ε, η συμβολή αυτού του δικτύου σε όλες μας τις σχολές και μεταξύ μας λέμε ότι πλέον δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε αν αυτού. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Καταρχάς, η ε, κατάρτιση στο ίδιο το Ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό, ε, την ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι πολύ σημαντική για τους δικαστές και νομικούς και θα έλεγα πως είναι γενικά εύκολο το να ε, εξοικειωθεί κανείς ε, με αυτό το δίκαιο, όμως το δύσκολο είναι να γνωριστεί με τις δικαστικές αρχές και να δικοδομηθεί, να δημιουργηθεί μια αμοιβαία εμπιστοσύνη και γι' αυτό αυτό το δίκτυο διαρκώς οδηγεί σε μια ανάμειξη, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας, από διάφορες εθνικότητες, ε, όπου βρισκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο σε πλαίσιο κοινών, ε, σε, κοινών ε, επαφών, σε, μέσω προγραμμάτων ανταλλαγών και αυτό βρίσκεται στην βάση αυτής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Δεύτερο παράδειγμα, Αρκετές χώρες, όλοι το γνωρίζουν, θυγήκαμε πολύ ε, σοβαρά από το, την τρομοκρατία και την βίαιη ριζοσπαστικοποίηση. Και χάρη στα δίκτυα αυτά, στους επόμενους αμέσως μήνες καταφέραμε να φτιάξουμε κοινή ε, κατάρτιση αλλά και ανταλλαγές για παράδειγμα για την κατανόηση αυτού του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης, την πρόληψη και το είδος των απαντήσεων και των προγραμμάτων από ριζοσπαστικοποίησης που μπορούσαμε να προβλέψουμε ή το πώς εξελίσσονται αυτά τα φαινόμενα σε συνθήκες κράτησης. Χάρη σε αυτά τα δίκτυα μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Ευρώπη, πράγμα ε, με αυτούς που είχαν περισσότερο θυγή ε, και να προσπαθήσουμε έτσι να εξοπλιστούμε καλύτερα και να κατανοήσουμε καλύτερα τα φαινόμενα αυτά. το παράδειγμα, διαφορετικό. Το γνωρίζετε, η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ε, σε όλες τις χώρες είναι ιδιαίτερα φορτωμένη. Η ζήτηση για δικαιοσύνη αυξάνεται, ενώ τα μέσα που αφιερώνονται δεν αυξάνονται ανάλογα και όλοι πρέπει να καταβάλουμε διοικητικού τύπου προσπάθειες. Ε, Γι' αυτό και οι πρόεδροι των δικαιοδοσιών και ε, οι εισαγγελείς έχουν και διοικητικό ρόλο να παίξουν και γι' αυτό χρειάζεται ε, να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε τις ε, καλύτερες πρακτικές και να υπάρχει έτσι μια ισορροπία αλλά και εγγύηση για ανεξαρτησία στην κάθε δικαιολογία. Πέρα από αυτές τις ε, συναλλαγές τις εξαιρετικά τεχνικές, ε, διαχέεται έτσι μια κοινή κουλτούρα για το τι πρέπει να είναι ένας οργανισμός ε, κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων και για τον ε, χώρο που καλύπτει από ε, αυτό το είδος οργανισμού μέσα στην θεσμική αρχιτεκτονική και σε ένα κράτος δικαίου. Και γι' αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από αίτημα των εθνικών σχολών, έχουμε καταλήξει σε κάποιες αρχές για την δικαστική κατάρτιση. Να σας τη συνοψίσω εν συντομία. Έχουμε κάποιες ε, αρκετά απλές ιδέες ως βάση, που όμως μας φάνηκε χρήσιμο να τις, να καταγράψουμε, τις βρίσκεται και στο έγγραφο που σας έχουμε δώσει. Καταρχάς, η ανάγκη κανείς να έχει περάσει από συγκεκριμένη κατάρτιση πριν να γίνει δικαστής ή εισαγγελέας. Είναι, φαίνεται προφανές, αλλά δεν είναι πάντα. Το να μάθει κανείς το δίκαιο δεν είναι μόνο μια θεωρητική ε, παιδεία, αλλά και μια πρακτική ε, παιδεία. Δεύτερη αρχή, δικαίωμα, μάλλον υποχρέωση να καταρτίζεται κανείς στη διάρκεια του επαγγελματικού του βίου γιατί εξελίσσονται οι ε, δικαστικές προδιαγραφές αλλά και οι τεχνικές επαγγελματικές εξελίσσονται και οι τεχνολογικές επίσης τεχνικές και έχουν πολύ έντονο αντίκτυπο στην δουλειά μας. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ε, και να μην περιορίζουμε αυτή την κατάρτιση, αυτή την, αυτού του είδους την εκπαίδευση στα, στη, γνώση του νόμου, του δικαίου. Δεν αρκεί αυτό. Το πώς γίνεται μια κροματική διαδικασία, ποια είναι η θέση του δικηγόρου, ποια είναι η στρατηγική για την διεξαγωγή μιας έρευνας. Όλα αυτά τα στοιχεία θεωρούμε πως είναι απαραίτητα και αποτελούν την καρδιά της επαγγελματικής κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων. Έχουμε λοιπόν σημαντική ευθύνη ώστε αυτή, η είδου η κατάρτιση να καταστεί δυνατή και υπό την ευθύνη των δικαστών και των εισαγγελέων είναι σημαντικό να τα εφαρμόζουν όλα αυτά και να μην τα εγκαταλείπουν. Το εξίσου είναι σημαντικό να συνδράμουν και οι ανώτατες δικαστικές αρχές, οι οργανώσεις πρόσληψης, κατάρτιση ε, του κλάδου ε, διαφέρουν, ε, αλλά εν πάση περιπτώσει το ανώτατο δικαστήριο όριο λόγος κάθε χώρας ε, στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την κατάρτιση. Τώρα, ποιες προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ένα που το γνωρίζετε είναι ο φόρτος εργασίας των δικαστών και εισαγγελέων ε, και αυτή, αυτός ο φόρτος έχει άμεσο αντίκτυπο για την κατάρτιση που ε, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν οι ίδιοι είτε από μόνο τους είτε υπό την πίεση των ιεραρχικά ανωτέρων τους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλα τα θέματα. Αυτή την ένταση τη γνωρίζουμε, τη ζούμε όλοι, είμαστε όλοι και εισαγγελείς και ε, ερχόμαστε από κάποιες δικαιοδοσίες, θα επανέλθουμε εκεί και ε, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να εντάξουμε το χρόνο κατάρτισης μέσα στην επαγγελματική μας πορεία. Φαντάζεστε βέβαια ότι για να οικοδομηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη πρέπει να μπορούμε να επικοινωνούμε εύκολα. Και γνωρίζετε καλά εδώ ποιες είναι οι προκλήσεις ε, όσον αφορά τις γλωσσικές ε, δεξιότητες. Συχνά προσφέρονται ε, μαθήματα γλωσσών, αλλά αυτά δεν αρκούν. Εργαζόμαστε πολύ επί τις ορολογίες, γιατί γνωρίζετε έχουμε και εμείς μια γλώσσα η οποία δεν είναι πάντοτε πολύ προσβάσιμη, αλλά τουλάχιστον τουλάχιστον μεταξύ μα πρέπει να μπορούμε να συνεννοηθούμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ συχνά το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι πιο καλά προσαρμοσμένο για να διευκολυνθεί η επικοινωνία και βεβαίω ε, αυτή την ευρωπαϊκή γλώσσα πρέπει να την μεταφράσουμε σε μια γλώσσα που να είναι κατανοητή από όλους τους ε, ε, τα 11 μέρη. Πρέπει να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα μέτρα λιτότητας σε διάφορες χώρες έχουν πλήξει και τις δικαστικές αρχές και αποτελούν τεράστια πρόκληση. Ε, Επίση θέλω να επιμείνω για τις νέες ανάγκες. Σας είπα ότι δεν πρόκειται μόνο για την κατάρτιση όσον αφορά το ίδιο το δίκαιο, αλλά γνωρίζουμε πως οι ανάγκες κατάρτισης υπάρχουν για τη διοντολογία, για την στάση, για την επικοινωνία με το σύνολο των πολιτών και των δίκων μερών και είναι πολύ σημαντικά αυτά και πρέπει να τα συζητάμε και το καταλαβαίνουμε ότι είναι εξίσου σημαντικά και τους Ευρωπαίους συναδέλφους. Επίσης, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που αντιμετωπίζουν νέες μεθοδολογίες εκμάθησης μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης ε, ή της εξαποστάσεως μάθησης μέσω του ίντερνετ, αλλά γνωρίζουμε πως υπάρχουν και περιορισμοί ε, στα μέσα αυτά και από αυτή την άποψη η ανταλλαγή ε, εμπειριών είναι πολύ χρήσιμη. Να σας πω ότι το δίκτυο αυτό λοιπόν που υπάρχει εδώ και 15 χρόνια έχουμε ξεκινήσει ένα προβληματισμό για το επόμενό μας στρατηγικό πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο, μάλλον για το οποίο τροφοδοτεί μάλλον αυτός ο προγραμματισμός στις δραστηριότητε μας και αυτό το στρατηγικό σχέδιο θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο ε, συντονισμένοι με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εξαρτώμεθα πολύ από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε μεγάλο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το, το στρατηγικό μας πρόγραμμα θα πρέπει να υιοθετηθεί για το 2020. Έχουμε μια διάσκεψη των διευθυντών όλων των σχολών τον φθινόπωρο του 2018 και τώρα ξεκινάμε τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι πολύ θα θέλαμε να μπορούμε μαζί σας να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτούς τους προσανατολισμούς, τις ε, ανάγκες που εσείς, που εσείς εντοπίζετε και το πώς θα πρέπει να ενεργήσουμε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισήγησή σας. Έχουμε κάποια λεπτά για ερωτήσεις από πλευράς των μελών. Ο κύριος Λεμπρετό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Δικτύου ε, Δικανικής εκπαίδευση μα δώσατε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και ευχαριστώ κυρίω την κυρία Σαγκάν που ήρθε και που μίλησε στα γαλλικά. Ε, πράγμα το οποίο σπανίζει. Η γλώσσα του Μολιέρου θα έπρεπε να αντυχεί πολύ περισσότερο εδώ σε αυτέ τι αίθουσε. Ωστόσο, λυπούμε κάπω γιατί το έγγραφο που μα δώσατε είναι συντεταγμένο μόνο στα αγγλικά και αποκλειστικό. γιατί από ό,τι κατάλαβα έχετε 10 εκατομμύρια ευρώ προπολογισμό. τέλο πάντων είναι πρότασή μου αυτή να χρησιμοποιήσετε ένα κομματάκι για να το μεταφράσετε από το κείμενο και στι άλλε κύριε γλώσσε τη Ένωση. Ε, ε, είναι πολύ ενδιαφέρον ε, τα όσα λέγονται εδώ και αυτό το δίκτυο και που επιτρέπει μία συνεργασία ανάμεσα στις κρατικές ε, δικαιοδοσίες και εγώ στηρίζω πάντοτε την συνεργασία μεταξύ των κρατών. Η τα όσα αναφέρονται δεν είναι πολύ θετικά. Πρώτον, η γνώση για τις άλλες δικαιοδοσίες σε υποκανονικές συνθήκες λειτουργίας. Αυτό ανοίγει το μυαλό, το πνεύμα των δικαστών μας και τους επιτρέπει να διαπιστώσουν τις καλές πρακτικές που υπάρχουν ε, στο εξωτερικό και έπειτα δεύτερο όφελος είναι το να μάθουν μεταξύ τους οι δικαστές να εμπιστεύονται αλλήλους, πράγμα που θεωρώ πολύ σημαντικό. Ε, τώρα, Υπάρχει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι κάπως ε, προβληματικό και ακατανόητο είναι ότι σχεδόν όλες οι ανταλλαγές δικαστών στην Ευρώπη γίνονται υπό την αιγίδα αυτού του δικτύου. Όμως υπάρχει και μια εξαίρεση ότι δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό διόλο μελιτέο ανταλλαγών που γίνεται εκτός ε, του πλαισίου αυτού, του δικτύου αυτού. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι είναι αυτές οι ε, ανταλλαγές και πώς οργανώνονται. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί να προσθέσω ότι δεν είμαι υπέρ των μονοπωλίων σε κανέναν ε, τομέα και ιδιαίτερα στον τομέα της ε, ε, κατάρτισης, της επαγγελματικής κατάρτισης είναι καλό να υπάρχουν διάφορες δυνατότητες. Ευχαριστώ. Ο κύριος ναι, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα διαμαρτυρηθώ εναντίον του ε, δικαστή Ποστόσκη διότι πραγματικά δεν μίλησε τα πολωνικά που είναι η όμορφη αυτή η γλώσσα η ωραία τόσο γλώσσα του Πάπα Βοητήλα και του Άντα Μίνιτς. Ε, πάντως ε, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση την οποία κάνατε. Ε, σας γνωρίζω κύριε δικαστά, συναντώμεθα κάπου κάπου. E, e, Νομίζω ότι αυτό το οποίο μου έρχεται στο νου είναι το εξής. Ίσως η ερώτησή μου δεν είναι τόσο σημαντική και ανοίξει νέους ορίζοντες, αλλά αναφερθήκατε σε διαφορετικές μορφές κατάρτισης, σημαντικές για τους δικαστές και σημαντικές για την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Ένωση. Μήπως θα ήταν δυνατόν τις προτάσεις σας να μας τις παρουσιάσετε κάπως πιο αναλυτικά σε σχέση με τα κέντρα εκπαίδευσης των στελεχών της δικαιοσύνης. μπορούμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία ε, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κέντρα αυτά, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα στενότερων σχέσεων των κέντρων και μεταξύ τους και με τα πανεπιστήμια και τις νομικές σχολές. Ο κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ μια απλή ερώτηση. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε ζήσει τρομερές τραγωδίες για τις οποίες δεν ήταν προετοιμασμένη η αστυνομία και το δικαστικό σώμα, η διεθνής τρομοκρατία τρέχει πιο γρήγορα και από το διεθνές έγκλημα κάτι το οποίο είχαν θέσει ήδη από το 2016 στις αρχές ο δικαστής Μπερτόσα και οι δικαστές και οι εισαγγελείς της Γενέβης. Τι λείπει λοιπόν σήμερα στην δικαιοσύνη, στους ανακριτές, έτσι ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν με υψηλότερη ταχύτητα και να μπορέσουν να προλάβουν ή έστω να συλλάβουν τους δολοφόνους και γιατί η τρομοκρατία στην Ευρώπη δεν είναι εθνική, είναι διεθνής. Είπατε ότι η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη, είναι αλήθεια, αλλά από την άλλη είναι ένα προϊόν το οποίο απαιτεί πάρα πολλά χρόνια για να εγκατασταθεί στις νοοτροπίες. Μήπως οι συνεργασίες αντιμετωπίζουν εθνικά εμπόδια τα οποία Οφελούν τους εγκληματίες. Ενθυμούμε ότι πολλά οφείλουμε στον κύριο Κάνιβεκ, ο οποίος εδώ ήταν αυτός που είχε ζητήσει να δημιουργηθεί το πρώτο δίκτυο των ανωτάτων δικαστηρίων. Σήμερα ε, το διεθνές χαρακτηριστικό της εγκληματικής δραστηριότητας ε, μήπως ε, έχει αν θέλετε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανημένες οι εθνικές δικαιοδοσίες. Κύριος Μαρίνιο. Ευχαριστώ. Εγώ άκουσα με πολύ προσοχή τα όσα μας είπατε και χαιρετίζω την ύπαρξη αυτού του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την επαγγελματική κατάρτιση των δικαστών. Έχω την εντύπωση ότι λείπει μία, ένας πυλώνας από αυτή την κατάρτιση και είναι η κατάρτιση των, των ε, των δικηγόρων. Επειδή είναι ελεύθερο επάγγελμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και, η Ευρωπαϊκή, και, και τα ευρωπαϊκά κράτη θα έπρεπε να ανησυχούν εξίσου για την κατάρτιση των δικηγόρων, γιατί αυτό το σύστημα το δικαστικό θα ζητήσει, θα λειτουργήσει σωστά μόνο εάν είναι καλοί οι δικηγόροι που είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτού του συστήματος. Γι' αυτό και νομίζω πως μια, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επαγγελματικής κατάρτισης, δικαστικής κατάρτισης θα έπρεπε να δώσει και μια προσοχή και στους δικηγόρους και την κατάρτιση αυτών. Τα εθνικά κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενδιαφέρονται το ίδιο για την ύπαρξη των καλών εισαγγελίων όπως και για την ε, ύπαρξη των καλών δικηγόρων. Και ανεξάρτητα από την κατάρτιση των δικηγόρων μέσω των δικών τους ενώσεων ε, ε, τα κράτη, τα έθνη, τα ευρωπαϊκά θα έπρεπε να αναλάβουν κάποια ευθύνη. Ιδιαίτερα με χρήματα, ώστε να μπορέσει να γίνει καλύτερη κατάρτιση των δικηγόρων που είναι όπως είπα αναπόσπαστο τμήμα του δικαστικού συστήματος κάθε χώρας. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω και την γνώμη των προσκεκλημένων μας ακριβώς για την ανάγκη καλών δικηγόρων για να μπορέσει όπως είπα να λειτουργεί ορθά το δικαστικό σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να λοιπόν αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Αν θα θέλατε να απαντήσετε σε όποια γλώσσα επιθυμείτε. Ε, επιτρέπω και την χρήση της γλώσσας του Σακεσπύρου, αλλά κατ' εξαίρεση μόνο. Ευχαριστώ. Πρώτα στα αγγλικά λοιπόν και μετά στα γαλλικά. Χρησιμοποιούμε αυτές τις δύο γλώσσες, διότι είναι οι δύο ε, γλώσσες εργασίας του δικτύου μας, του JTN. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η προσφορά της εκπαιδεύσεως γίνεται μόνο σε αυτές τις δύο γλώσσες. Και όταν παράγουμε το σχετικό υλικό, όπως το εγχειρίδιο μεθοδολογίας του JTN, αυτό εκδόθηκε σε όλες τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και οι αρχές που ανέφερε πριν η Βαλερή, και αυτές είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης. Είναι βέβαια μεγάλο ο γλωσσικό πλούτο τη Ένωση. Οι εκπαιδεύσει μα δεν γίνονται μόνο σε γαλλικά, αγγλικά, αλλά και σε ισπανικά, γερμανικά και ιταλικά. Γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά. Αυτά κάνει το JTN και προσφέρει και τι αναγκαίε ε, και τις αναγκαίους πόρους χρηματοδοτικούς δηλαδή. Θα απαντήσω τώρα πρώτα για την ερώτηση για το πρόγραμμα ανταλλαγής Αυτό βέβαια κυριαρχεί στις ανταλλαγές που γίνονται στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα όπως τώρα δεν είναι πολύ μεγάλο. Στέλνουμε τους δικαστές για δύο εβδομάδες σε άλλη χώρα μέρος. Αυτό είναι το βασικό πρόγραμμα. Κάνουμε όμως και πιο ειδικευμένε ανταλλαγές για το ε, δίκαιο του ασύλου, για το δίκαιο του περιβάλλοντος, για το δίκαιο ε, για μελλοντικούς, ε, μάλλον εκπαιδευόμενους δικαστές που τους στέλνουμε σε άλλες χώρες μέλη. Στέλνουμε δικαστές και σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στα δικαστήρια, στο Στρασβούργο. Και το πρόγραμμά μας κυριαρχεί στις ανταλλαγές δικαστών, χωρίς να έχουμε βέβαια το μονοπόλιο. Γίνονται κάποιες μικρότερες ανταλλαγές, όπως και για τα ανώτατα δικαστήρια που οργανώνονται από άλλους φορείς στην Ευρώπη. Όμως η οργάνωση των ανταλλαγών είναι τεράστια πρόκληση. Το JTN θεσπίζει κανόνες. Δεν είναι βέβαια πολύ μεγάλο το βάρος που επιβάλλουμε στις εθνικές αρχές. Από άλλα θεσμικά όργανα προσπαθούν, είναι δύσκολο βέβαια να εντοπιστούν οι συνάδελφοι και να συνδυαστούν και τα εκπαιδευτικά τους ενδιαφέροντα αλλά και οι γλώσσες που μιλούν κτλ. Χρειάζεται και μεγάλη εμπειρία. Γι' αυτό φαίνεται σαν το δίκτυό μας να μονοπολεί τον με αυτό. Όμως προσπαθούμε ε, να ανταποκριθούμε σε όλες τις ανάγκες που εντοπίζονται. Η οργάνωση είναι καλή για τους δικαστές. Σύμφωνο. ότι θα πρέπει να αρχίσουμε, ε, να αρχίσουμε να επενδύουμε στους νέους ανθρώπους όταν αρχίζουν να μελετούν τις σταδιοδρομίες τους ε, στο δικαστικό σώμα. Γι' αυτό το JTN αποδίδει μεγάλη σημασία στους εκπαιδευμένους, στους ασκουμένους, αυτοί δηλαδή, αυτούς δηλαδή που αρχίζουν όταν έχουν πάρει το πτυχίο τους από την νομική σχολή δεν έχουν ακόμα όμως διοριστεί δικαστές, εισαγγελίες κτλ. Έχουμε και το πρόγραμμα Ζάκος, το οποίο είναι πρόγραμμα ανταλλαγή ασκουμένων για να ανοίξει το πνεύμα τους στο ευρωπαϊκό δίκαιο με τρόπο διαφορετικό από αυτό που κάνουν τα πανεπιστήμια τους. Έχουν και διαγωνισμούς όπου διαγωνίζονται οι ε, νέοι ασκούμενοι για να αποδείξουν το επίπεδο των γνώσεών τους στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Έχουμε τώρα και θερινά σχολεία με εξειδικευμένη εκπαίδευση για τους ε, ασκουμένους αυτούς. Δεν συνεργαζόμαστε τόσο με τα πανεπιστήμια. Θεωρούμε ότι η δική μας εκπαίδευση είναι διαφορετική από αυτήν των πανεπιστημίων, αν και έχουμε πολλούς πανεπιστημιακούς οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μας. Όμως η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε εμείς είναι στοχευμένη σε επαγγελματίες, δηλαδή σε ε, ενηλίκους οι οποίοι είναι ήδη επαγγελματίες, είναι αρχίζουν, δηλαδή είναι ήδη ασκούμενοι. Είναι διαφορετικό από αυτό που προσφέρεται στους φοιτητές. Δεν λησμονούμε όμως το πανεπιστημιακό επίπεδο και εποφελούμεθα και από τις γνώσεις τους. Όταν μιλούμε για τα διαφορετικά επαγγέλματα, συμφωνώ ότι η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος δεν βασίζεται μόνο στους δικαστές και εισαγγελείς, αλλά και στους δικηγόρους, ε, δικαστικούς γραμματείς, ε, δικαστικούς επιμελητές και ούτω καθεξής, οι οποίοι όλοι αυτοί πρέπει να είναι ορθά εκπαιδευμένοι. Στο GTN, καθήκον μας, αποστολή μας είναι να εκπαιδεύουμε δικαστές και εισαγγελείς, αλλά δεν είμαστε κλειστοί σε αυτό. Συνεργόμαστε ε, στενά και με το CCB, την Ένωση δηλαδή των Δικηγορικών Συλλόγων στην Ένωση και αναζητούμε και τρόπους συνεκπαίδευσης αν και δεν είναι δικό μας καθήκον αυτό, δηλαδή να εκπαιδεύονται ταυτόχρονα δικαστές εγγελίσεις και δικηγόροι. Ούτε είναι και τόσο εύκολο να, συνεργα... να ε, οργανωθεί η εκπαίδευση των δικηγόρων στο ίδιο επίπεδο όπως για δικαστές και αγγελίε, γιατί εμείς βρισκόμαστε στην πιο άνετη θέση όλες οι χώρες μέλη να έχουν δημόσιους θεσμούς οι οποίοι να εκπαιδεύουν δικαστές και εισαγγελείς. Ενώ οι δικηγόροι εκπαιδεύονται από τους εθνικούς δικηγορικούς συλλόγους. Άρα η σχετική δικτύωσή τους γίνεται πιο δύσκολη. Όπως είπα, το JTN προσπαθεί να εντοπίσει πού βρίσκονται οι ανάγκες για κοινή εκπαίδευση. Και όπως είπα, κάνουμε κάποιε κοινέ εκπαιδεύσει με τους δικηγόρου το ίδιο με αστυνομικούς ε, ε, διευθυντές κτλ. Βεβαίω αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται προσεκτικά. Μη λησμονούμε ότι οι δικαστέ είναι ανεξάρτητοι και τους αρέσει να, έχουν ένα, ε, να μπορούν να εκπαιδεύονται σε ένα περιβάλλον ασφαλές όπου να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις απολύτως ελεύθερα. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε ευγνώμονε για την γεωνοδορία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, η κατάσταση έτσι έχει ω τώρα. Δικαστέ και εισαγγελεί είναι εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν την πλουσιότερη εκπαιδευτική προσφορά στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ και να μου επιτρέψετε να παραδώσω το μικρόφωνο στη συνάδελφή μου Βαλερή. Για να συμπληρώσω λίγο για το θέμα των ανταλλαγών εκτός δικτύου. Euh, euh, Πράγματι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες ανταλλαγών που βασίζονται είτε σε προσωπικές σχέσεις ή σε κάποια πολύ πιο διεθνικά συστήματα που αφορούν πολύ περισσότερες σε πολύ περισσότερες από α, λίγες χώρες. Εμείς δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα μονοπωλιακά. Σε επίπεδο διακυβέρνησης δεν υπάρχει μια υπερδομή η οποία να μας κατευθύνει όλους. Έχουμε μια χαλαρή δομή η οποία εκπροσωπείται από τη γραμματεία και η οποία μας βοηθά σε πρακτικό επίπεδο διευκολύνοντας τις επαφές. Γιατί καταλαβαίνετε ότι σε επίπεδο διαδικαστικό πολλές φορές είναι απαιτητικά τα πράγματα. Δεύτερον, για τους δικαστές και εισαγγελείς πριν από το διορισμό τους. Επανέρχομαι σε αυτά τα οποία είπε ο Βόιτσεκ. Είναι ένα από τα θέματα που έχουμε μπροστά μας, το επόμενο στρατηγικό πλάνο μας, να παρέχουμε ακόμα περισσότερες δυνατότητες σε αυτούς που ξεκινούν την επαγγελματική τους καριέρα. Γιατί τη δική σας ερώτηση, Πρόεδρε, εγώ δεν έχω την δυνατότητα ούτε την εντολή να απαντήσω με επακριβή τρόπο και δεν μπορώ να σας δώσω μια επακριβέστατη εικόνα ενός θέματος που ξεπερνά κατά πολύ τα θέματα της κατάρτισης. Μπορώ να σας μεταφέρω μια αντίληψη περισσότερο που έχω ότι σε σχέση ιδιαίτερα με τη συνεργασία σε ποινικό ε, επίπεδο και για την ε, τρομοκρατία ε, οι δικαστές και οι εισαγγελείς εκτιμούν τα κοινά μέσα. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψη σαφώς και έχει βοηθήσει τα πράγματα και το Eurojust βοηθά πολύ, αλλά θα μπορέσει ίσως να βοηθήσει και περισσότερο εάν οι ικανότητες οι οποίες έχουν αποδοθεί στο Eurojust αναπτυχθούν έτσι περαιτέρω. Ε, συνειδητοποιούμε αυτή τη δυτή κίνηση, μια κίνηση αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης. Ξέρετε ότι το ποινικό είναι περίπλοκο δίκαιο και γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε να καταστεί ή να καταστούν οι διάφορες μορφές απόδοσης ή ερμηνείας του ποινικού δικαίου με τρόπο ε, μεταξύ τους συμβατές. Κάτι το οποίο θα προωθήσει με λειτουργικό τρόπο την συνεργασία. Πάντως έχουμε ανάγκη από διάφορα μέσα συγκεκριμένα έτσι ώστε να θεσμοποιηθεί αν θέλετε η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω διαδραστικότητας ανάμεσα στους εμπλεκομένους. Ε, πάντως εγώ δεν έχω κάποια ιδιαίτερη επαϊοσύνη επί του συνολικού θέματος, αλλά κάποιες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ανταλλαγές ανάμεσα σε επαγγελματίες του δικαστικού σώματος. Σας ευχαριστώ και τους δύο ομιλητές που ήρθατε εδώ μαζί μας και μας ενημερώσατε. Τελειώσαμε λοιπόν το δημόσιο τμήμα της συνεδριασής μας για σήμερα. Η συνεδρίαση θα συνεχιστεί και κλεισμένων των θυρών. Ιωσδήποτε δεν δικαιούται να συμμετέχει παρακαλώ να εγκαταλείψει τον χώρο.